Goed, collega's. Ik stel voor dat we. προτείνω να προχωρήσουμε για όσους δεν ήσαν παρόντες να πω πως ε, ψηφίσαμε για την υποψηφία του κυρίου Λέινα 17 ψήφοι υπέρ, 4 κατά και 2 αποχές ήταν το αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, κυρία Γιάλας γνωρίζει τι θα συμπεριλάβει στην εκθεσή της. Περνάμε στο επόμενο σημείο, σημείο 5, απαλλαγή για το 2012, σκηνές επιχειρήσεις. Ο κύριος Ρούμπιχ είναι εισηγητής, αλλά μου είπαν ότι αυτή τη στιγμή ψηφίζει στην Επιτροπή Ήτρε και η κυρία Γκρέσλερ θα τον αντικαταστήσει. και αν φτάσει εγκαίρος τότε θα συνεχίσει ο κύριος Ρούμπιχ. Δώσω το λόγο καταρχήν στο ελεγκτικό συνέδριο. Έχουμε δύο εκπροσώπους. Το ελεγκτικό συνέδριο, τον πρόεδρο Μάρκ Κρίστο, τον διευθυντή Μάρκ και τον κεφαλής ε, ε, ε μονάδας Μπέρτραν Αλμπίγκ. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Καλημέρα σας. Όπως γνωρίζετε, η εντολή του Ελληνικού Συνεδρίου είναι να εκδίδει γνωμοδοτήσεις, μία για το ζήτημα της, των, των συναλλαγών και μία για τις δραστηριότητε. Το 2012 συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι υποδείξεις για τέσσερις τομείς, ε, για ε, εσωτερικό έλεγχο, παρακολούθηση και θέματα ε, πνευματικής διοκτησίας. Για πρώτη φορά λοιπόν ε, υποβάλαμε μια συνοπτική έκθεση. Είναι ένα σημαντικό έγγραφο για αυτό το οποίο συντάσσουμε ετησίως για τις επιχειρήσεις όπου συμπεριλαμβάνονται οι παρατηρήσεις μας για όλες τις κοινές επιχειρήσεις. Τώρα κάνουμε διάφορες αναλύσεις, αξιολογήσεις, έλεγχο των συστημάτων και το θέμα των ε, συναλλαγών. Ε, το ε, ex έλεγχος είναι θέμα κλειδί για τις εξελίξεις το θέμα των ε, σε ό,τι φορά την νομιμότητα και την ε, μη νομιμότητα της παρατυπής ε, διάφορα ζητήματα FCA, FCH, CSR, Clean Skies κλπ. Εκδώσαμε λοιπόν τρεις ε, νομοθετήσεις για την IMI, Innovative Medicines και Επίσης, σε ό,τι φορά το ανάρθεμι και την ENIAC, οι προφορίες που ήταν διαθέσιμες για την εφαρμογή του έξπος του ελέγχου δεν επάρκησαν προκειμένου να καταλήξουμε ότι το ζήτημα αυτό η ε, έλεγχο λειτουργήσε αποτελεσματικά. Κάναμε και παρατηρήσεις που είναι σημαντικές, αλλά όχι απαραίτητο να επηρεάζουν τη γνώμη της, ε, του Συμβουλίου ότι δηλαδή έχουν, ε, υπολείπονται κατά 50% οι, οι πληρωμές πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των διαδικασιών των προμηθειών, ο εσωτερικός έλεγχος της Επιτροπής και των κοινών επιχειρήσεων που υιοθέτησαν μικτές αυτές επιχειρήσεις ε, όπως η Artemis, η σενία και η ΚΑΠΑΦΗ δεν τροποποιήθηκαν για να συμπεριλάβουν ε, τις αλλαγές ε, που προέκυψαν. Και τέλος το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, το FP7, καθορίζει ένα σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου οι περισσότερε ε, τις θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω αυτέ τι ε, υποδείξει. Ε, θα θέλαμε να κάνουμε κάποιε συγκεκριμένε παρατηρήσει αναφορικά με το θέμα τη σύνδεξη για το πρόγραμμα Ίντερ και με την προσοχή στο θέμα του κόστου στο ζήτημα τη κατασκευή του Ίντερ. Το ποσό ήταν 6,1 δις δολάρια αλλά ε, έχουμε, ε, ε, τα προκύπτει ότι θα υπάρξει παρέκκληση από αυτό το ποσό. Κατά 290 εκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και μέλη του Επιστατού του Ελέγχου Προπολισμού. Είμαστε να, να απαντήσουμε σε συγκεκριμένε ερωτήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει ο συνάδελφος το λόγο μήπω από το ελεκτικό συνέδριο. Κυρία Γκρέσλε, θέλετε να πάρετε το λόγο ή να δώσω το λόγο κατευθείαν στις κοινέ επιχειρήσεις. Κυρία Γκρέσλε, ίσως οι κοινέ επιχειρήσεις πρώτα. Λοιπόν, οπότε, να ακούσουμε τους παρόντες, τους εκπροσώπους από τις κοινέ επιχειρήσεις που κάθεστε... Α, από εδώ. Συγγνώμη, συγγνώμη, η περιφερειακή μου όραση λίγο πάσχει. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα αριστερά προ τα δεξιά. Έτσι. Ποιο θέλει να μιλήσει πρώτο, Παρακαλώ. Ε, πείτε μα εσείς από ποια, κοινή επιχείρηση εκπροσωπείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μιλήστε καλύτερα στο αριστερό μικρόφωνο, είναι καλύτερα για σας. Ευχαριστώ. Είμαι ο εκτελεστικός διευθυντής ε, της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα του IMI και θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας το Ελεκτικό Συνέδριο γιατί βλέπω ότι μετά από 4,5 χρόνια δραστηριοτήτων έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο ρήμανσης και οι ε, εκθέσεις του ε, συνεδρίου μας βοηθούν πολύ για να προχωρήσουμε θα επικεντρωθώ σε αυτή την σύντομη δήλωσή μου μόνο στο βαθμό λάθους, που είναι περίπου στο 2% που είναι το όριο για την ε, έγκριση των εκθέσεων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το θέμα αυτό το διερεύνησε και το δικό μας εσωτερικό σύστημα ελέγχου πριν γίνει παρατήρηση από το ελεγκτικό συνέδριο που νομίζω ότι δείχνει και την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του δικού μας εσωτερικού συστήματος ελέγχου. Ποια είναι τώρα, ποιος είναι ο λόγος μάλλον γι' αυτό. Γιατί θα μπορούσατε να πείτε, αφού το βρήκατε το λάθος, γιατί δεν το διορθώσατε. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Καταρχάς, το είδος των δικαιούχων. Εμείς έχουμε να κάνουμε με δικαιούχους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Ξέρετε ότι οι μεγάλες εταιρείε γνωρίζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αλλά δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω του IMI. Από την άλλη όμως προσελκύουμε πολλές ακαδημαϊκές ε, ομάδες ε, καινοτομίας, ε, από παντού, από όλε τι χώρες τη Ευρώπης, οι οποίε όμως δεν είναι απολύτως εξοικειωμένε με, το, με τα ευρωπαϊκό Οπότε, τι κάναμε για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Πήραμε κάποια μέτρα έτσι ώστε να, ε, να μειώσουμε τον, ε, τον βαθμό λάθους. Για παράδειγμα, υποβάλαμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στους δικαιούχους, τις οποίες ενημερώνουμε τακτικά. Ε, αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές ε, τους ε, παρουσιάσαμε και σε συγκεκριμένα εργαστήρια. Κάναμε πολλούς, πάνω από 100 ελέγχους και πήραμε κάποια μέτρα για να εφαρμόσουμε την ανάκληση των αχρεωσίδων καταπληθέντων ποσών. Και βεβαίω προσπαθήσαμε να δούμε τι γίνεται και με του εξάντε ελέγχου. Αυτό λοιπόν που θέλαμε να δούμε είναι ε, τα συστήματά μα να μπορούν να ε, δίνουν αυτόματα εκθέσει για να μειώνεται ο βαθμό λάθου. Νομίζω ότι αυτό ήταν αρκετά αποτελεσματικό γιατί έτσι με τα μέτρα αυτά μειώσαμε το βαθμό λάθου στο επίπεδο του 3,6%. Οπότε, αυτό που θέλω να πω, κλείνοντας, είναι ότι ε, παραμένουμε αφοσιωμένοι στη διαχείριση ε, της χρηματοδότησης, ε, έχοντας υπόψη ότι θα πρέπει βεβαίως να, γίνεται, ε, να υπάρχει έλεγχος αλλά και λογιστικός έλεγχος ενημερώνουμε το προσωπικό μας έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρησιμοποιούνται χρηστά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στον τομέα της υγείας αυτό σημαίνει ε, δημιουργία νέων ε, θεραπείων και για τις διάφορες ασθένειες. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι πέρσι καταφέραμε να δεσμεύσουμε όλον τον προπολογισμό, να εκτελέσουμε όλον τον προπολογισμό που είχε δοθεί στο IMI1. Πετύχαμε πάνω από 99% εκτέλεση προπολογισμού και σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις και τις πληρωμές. Το νέο project που έχουμε ξεκινήσει, το νέο πρόγραμμα, ε, είναι πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσει αρχές του έτους ένα ε, project που θα αφοσιωθεί στο Alzheimer με 14 φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες συμφώνησαν να συνεργαστούν σε συνεργασία με, ε, οργα... με ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με τον ακαδημαϊκό κόσμο για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση. Και έχουμε κάνει ε, επίσης μεγάλη πρόοδο και στην αντιμικροβιακή αντίσταση. Οπότε, νομίζω ότι γενικώς το IMI προχωράει ε, και γίνεται η ναυαρχίδα της Ευρώπης στον τομέα της ε, υγείας και πρέπει να σας πω ότι και παντού στον κόσμο, κυρίως της ΕΠΑ, ε, προσπαθούν να αναπαράγουν αυτά που κάνουμε εμείς. Μας βλέπουν και μας μιμούνται. Αυτά που κάνουμε εμείς βέβαια με τη δική σας βοήθεια και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τη στήριξη σας αυτή και για τα επόμενα IMIs. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας. Σας ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Πάμε τώρα στον κύριο Ζενιό από την ΕΝΙΑΚ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μάρκ Ζενιό ονομάζομαι και εκπροσωπώ την ΕΝΙΑΚ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί ο εκτελεστικό μας διευθυντή, ε, ο κύριο Βίλκ, δεν μπόρεσε να, παρε, να παρίσταται σήμερα. Οπότε θα κάνω ό,τι μπορώ για να σα μεταφέρω το μήνυμα που μου ζήτησε. Καταρχάς θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το τι έχει γίνει τελευταίως στην ΕΝΙΑΚ. Διότι έληξε το πρόγραμμα πριν από μερικές εβδομάδες και με χαρά σας ενημερώνω ότι αξιοποιήσαμε 94% του προϋπολογισμού που είχε δοθεί στην ε, οργάνωσή μας. Επιλέξαμε 63 προγράμματα και Επίσης ε, ε, δεν ε, δαπανίσαμε όλα όσα προβλέπονταν για, τα λειτουργικά, για τις λειτουργικές δαπάνες. Όλα αυτά που δαπανίσαμε μόχλευσαν 2,9 δις επιλεξίμων δαπανών. Αυτό είναι κάτι το οποίο καλωσόρισαν και τα κράτη-μέλη και οι κλάδοι που συμμετέχουν στην ΕΝΙΑΚ. Ποιοι συμμετέχουν. Το τέλος αυτής της πρώτης φάσης, 24% μεγάλες εταιρείες, 45% μικρομεσαίες και 31% πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα. Αυτά είναι τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Τώρα για την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. λάβαμε υπόψη πολύ σοβαρά την ε, έκθεση του συνεδρίου για τον εκ των έλεγχο. Υπήρχε τριμερής ε, συμμετοχή και από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη. 23 κράτη-μέλη συμμετέχουν στην ΕΝΙΑΚΑ και φυσικά και ο κλάδος. Είναι λοιπόν ε, πολύ ε, εκτεταμένη η συμμετοχή και υπήρξε εκ των υστέρων έλεγχος γιατί οι δικές μας ε, οι εφαρμογές σε ό,τι αφορά την ε, χρήση του προπολογισμού από τα κρατημέλη σημαίνουν ότι ε, θα, ε, θα υπάρξει έλεγχος σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες. 23 διαφορετικές δέσμες κανόνων μιλάμε τώρα. Βεβαίως μιλάμε για πολύ περισσότερα χρήματα από όσα μπαίνουν στο πρόγραμμα και αυτή ήταν η επιλογή που τελικά ε, θεωρήσαμε ότι είναι η πιο σωστή. Πέρσι, από το 2012, ε, πέραν ε, αυτής της δραστηριότητας, κάναμε αρκετούς ελέγχους και δοκιμές και πέρσι δημιουργήσαμε ένα, καταρτήσαμε μάλλον ένα δείγμα με 161 συναλλαγές, με επικοινωνία με τα κρατη για τον συγκεκριμένο έλεγχο. Επίσης, έχουμε κάνει μια αξιολόγηση όλων των πιστοποιητικών που έχουν ε, κοινοποιηθεί από τις εθνικές αρχές Έχουμε λοιπόν μια διαδικασία που κινούμε τα κρατημέλη για να ελέγχουμε την ε, ε, πιστότητα, των, ε, την, το κατά πόσο είναι πρωτότυπα τα πιστοποιητικά. Και μπορούμε να εκδώσουμε και κατευθυντήρες γραμμές για να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση με τα κράτη-μέλη. Αυτά, Πρόεδρε, εδώ βρισκόμαστε. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει με τους ex post ελέγχους. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Φώστερ από το Artemis. Πρόεδρε, καταρχάς να ευχαριστήσω το Ελληνικό Συνέδριο για αυτή τη ε, διαδικασία. σω να είναι παράξενο, αλλά η συνεργασία μαζί, μας, μαζί τους μας βοήθησε να δημιουργήσουμε έναν πολύ πολύπλοκο μηχανισμό όλα αυτά τα χρόνια, με ένα μοντέλο τριμερούς χρηματοδότησης. Κατανοούμε βεβαίω ε, πολύ καλά τις ανησυχίες που έχει το Ελληνικό Συνέδριο για τους εξπόστα ελέγχου αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για την χρηματοδότηση και για να βρούμε ένα, μια προσέγγιση που θα συνάδει και με την επικουρικότητα, γιατί και τα κράτη-μέλη έχουν το δικό τους, τη δική τους ευθύνη στον όλο έλεγχο. Βεβαίως πρέπει να σεβόμαστε τα όσα ορίζει ο, ο κανονισμός του Συμβουλίου, οπότε τώρα προσπαθούμε με το Ελεκτικό Συνέδριο να βρούμε έναν συμβιβασμό, ο οποίος θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε σε ό,τι ε, αφορά τις δραστηριότητές μας. Είχαμε το προνόμιο να εργαστούμε σε αυτό το περιβάλλον και να συγκεράσουμε όλες αυτές τις, όλους αυτούς τους διαφορετικούς πολιτισμούς. Βεβαίως πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Επίση, λάβαμε κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όταν ένα σχέδιο υποβάλλεται, και μάλιστα είχαμε τις, όταν δημιουργήθηκε η δική μα κοινή επιχείρηση το 2008, δεν ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτή την τεράστια οικονομική κρίση που είχε να κάνει με τεράστια μέτρα λιτότητα και βεβαίω περιόρισε πάρα πολύ την συμμετοχή των κρατών μελών. Θυμόμενοι βέβαια ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτό που δίδεται από τα κράτη-μέλη, ε, βρεθήκαμε στην, στο να πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια σημαντική ε, μείωση του προπολογισμού. Τούτου λεχθέντος, ε, στο τέλος του προγράμματος καταφέραμε να επενδύσουμε κάτι λίγο παραπάνω από ένα δις ευρώ σε διάφορες δραστηριότητε έρευνας και ανάπτυξης ε, που οδήγησαν σε ε, μεγάλα ωφέλη σε ό,τι αφορά την δυνατότητα καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε είναι οι καθυστερήσεις διάθεσης του προπολογισμού. Ε, στην αρχή δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε αυτό το 2008, όπως σας είπα, αλλά υπήρξαν κάποιες ασυμμετρίες στην όλη προσέγγιση ανά χώρα για την χρηματοδότηση που, είχε να κάνει με την που οδήγησε σε καθυστέρηση της εκτέλεσης του προπολογισμού. Και προσπαθούμε από κοινού με τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν να βρούμε πρακτικές λύσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα και σας ευχαριστώ πολύ. Ehm, eh, ευχαριστώ πολύ η κυρία Γκρένς που τον κύριο Ρούμπιχ. Α, α, έχει έρθει ο κύριο Ρούμπιχ εδώ μεταξύ. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Παρακαλώ. Παρακαλώ, είστε ο συγητής, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε, ήμουνα στην Ήτρα, όπου ψηφίζαμε για το ίδιο θέμα και στην Ήτρα συζητάμε για το μέλλον, αλλά και εδώ συζητάμε για το μέλλον. Γιατί είναι πολύ σημαντική η εξέταση αυτών που έχουμε κάνει. Ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο ιδιαιτέρως. Αλλά το ελεγκτικό συνέδριο βέβαια δεν υπεύθυνο για το αν έχουν ανέβει ε, τα ποσοστά σφάλματος. Κυρίως ε, πρέπει να παίξει ένα προληπτικό ρόλο για αυτές τις κοινέ επιχειρήσεις. Μας ενημέρωσε λοιπόν ούτω ώστε να διαμορφώσουμε στο μέλλον καλύτερα και με βάση την πείρα αυτά τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν τις ε, ε παρουσιάσεις για το ποστό σφαλμάτων. Αυτό είναι πολύ καλό. Και οι ίδιες οι κοινέ επιχειρήσεις ε, αναγνώρισαν την ανάγκη βελτίωσης, άρα θα έχουμε βελτίωση στο μέλλον. Έχουμε και νέες ε, βασικές προϋποθέσεις, ένα νέο πλαίσιο. Τονίζω ότι στόχος μας είναι οι πιστώσει υποχρεώσεων και πληρωμών στο μέλλον να βελτιωθούν, να βελτιωθεί δηλαδή η αξιοποίησή τους. Βεβαίως προσπαθούμε να αποφύγουμε τις περικοπές, αλλά φυσικά το βασικό είναι οι πιστώσεις να αξιοποιούνται, γιατί αν δεν αξιοποιούνται πλήρως, μετά έχουμε περισσότερες περικοπές εφόσον δεν αξιοποιούνται υπάρχουσες πιστώσεις. Όντως πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την κατάσταση και σε σχέση με τις προθεσμίες για την ε, κατανομή των ε, προγραμμάτων. Στον τομέα της έρευνας είναι πολύ σημαντικό αυτό να χορηγούνται εύκολα και γρήγορα οι χρηματοδοτήσεις γιατί ο χρόνος ε, για τέτοια προγράμματα είναι πολύ σημαντικός. Αυτό το γνωρίζουμε. Ευχαριστώ τους πάντες. Είμαι ικανοποιημένος ιδιαίτερα με τις κοινέ μας επιχειρήσεις. Θα βοηθήσουν ε, και στο μέλλον και ελπίζω το ποσοστό για την ε, βιομηχανία να ανέβει στο 20% και πιστεύω ότι χώρες όπως η Γαλλία και άλλες πρέπει οπωσδήποτε να καλύψουν την καθυστέρησή τους και επειδή βεβαίως δεν είναι παντού ε, άριστη η οικονομική κατάσταση Πρέπει να βοηθήσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί όπως ξέρουμε 80% των θέσεων εργασίας δημιουργούνται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ λοιπόν τις κοινέ επιχειρήσεις που δεν ξεχνάνε τις μικρομεσαίες και τις θέσεις εργασίας που δημιουργούν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο από πλευράς των συναδέλφων. Ποιος? Παρακαλώ, κύριο Σταυρακάκης. με βάση τις προηγούμενες επιχειρήσεις το συνέδριο λέει ότι ναι μεν οι κοινέ επιχειρήσεις έχουν επιτύχει πρόοδους πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά για το σχέδιο για την ε, αντιμετώπιση των ε, θεομηνιών. Τι μέτρα πήρε το δικαστήριο προς αυτή, το συνέδριο για αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, η αξιοποίηση των πιστώσεων είναι στο 50%. Τι βελτιώσει έχουμε το 2013. Και μία ερώτηση στην κοινή επιχείρηση ENIAC. Η χρήση των πιστώσεων πληρωμών ήταν 52% το 2012. Σε τι βαθμό βελτιώθηκε αυτό το 2013. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Λοιπόν, παρακαλώ να απαντήσει σε ερωτήσεις του κυρίου Σταυρακάκη για την ΕΝΙΑΚ. Η πρώτη ερώτηση. Μιλάτε για το σχέδιο για ανάκτηση από τις θεομήνιες είναι οριζόντια δραστηριότητα, στην οποία δουλεύουμε πάντα. Υπάρχουν ε, πέντε κοινέ επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτό. Υπάρχει μεγάλη πρόοδος τον τελευταίο χρόνο. Δεύτερη ερώτηση. Για το Άρτεμις, ποσοστό εκτέλεση του προπολογισμού. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στη στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να έχουμε τις αναγκαίες ε, συμμετοχές και μεταφορές στους ε, συμμετέχοντες. Θέλουμε οι διοικητικές διαδικασίες μεταξύ των κρατών μελών και της ε, κοινής επιχείρησης Άρτεμις να είναι όσο ταχύτερες ε, γίνονται. Έχουμε κάνει μια μικρή αλλά σημαντική οργανωτική αλλαγή. Έχουμε έναν συγκεκριμένο αρμόδιο. Αυτό έχει βελτιώσει την κατάσταση τον τελευταίο χρόνο. Έχει υπάρξει μεγάλη βελτίωση που έχει θετική επίπτωση και στο ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Απάντησα σε ερωτήσεις σας. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Από τους εκπροσώπους του Ελληνικού Συνεδρίου υπάρχει τίποτα. Ούτε ο κύριος Ρούμπιχ. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη συμμετοχή σας. Ήταν πολύ χρήσιμη. Άρα μπορούμε να ε, προσβλέπουμε στη χορήγηση απαλλαγής. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το θέμα και περνάμε στο επόμενο θέμα. Η συγκίτρια είναι η κυρία Κάλτινμπαχ. Πρόκειται για την ειδική έκθεση 2013, κοινή γεωρική πολιτική, οι ειδικέ ενισχύσεις με βάση το άρθρο 86 του κανονισμού. Έχουμε εδώ τον Edward Χένεση από το Ελεκτικό Συνέδριο Οπότε να στραφώ προς το ελεγκτικό συνέδριο. Κυρία Κάλτενμπαχ, να ακούσουμε πρώτα το ελεγκτικό συνέδριο. Βεβαίως, ο κύριος Χένεση. Ε, thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Ελεκτικού Συνεδρίου που δεν μπόρεσε ένα μέλος μας να είναι παρόν στην Επιτροπή για να σας ε, παρουσιάσει την έκθεση σήμερα. Σας διαβεβαιώ όμως ότι αυτό δεν έχει να κάνει με έλλειψη ενδιαφέροντος για την εργασία της Επιτροπής σας, ούτε για το πώς αντιμετωπίζει αυτή την ειδική έκθεση. Αυτό συνέβη απλώ γιατί όλα τα μέλη του ε, συνεδρίου πρέπει να είναι παρόντα για τη συνεδρίαση σήμερα για να εκλεγεί ο πρόεδρο. Στην διαποσία ε, του λοιπόν θα σα παρουσιάσω εγώ την έκθεση. Και κάνοντας το θα είμαι σύντομος γιατί η κυρία Κάντεμπαχ η συγγήτρια έχει πραγματικά ε, συνοψίσει εξαιρετικά το περιεχόμενο της έκθεσης στο έγγραφο εργασία της. Θα επικεντρωθώ λοιπόν σε κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία θέλει να παρουσιάσει το Ελληνικό Συνέδριο. Όπως ξέρετε, το ε, πρόγραμμα ενιαίων πληρωμών ε, υιοθετήθηκε το 2003 και βασίστηκε πάνω στις αρχές των, ε, ε, της αποσύνδεσης ε, άμεσων πληρωμών από την παραγωγή και έτσι στην απλούστευση του καθεστώτος πληρωμών για, για τη Γεωργία. Ε, ως παρέκκληση από αυτές τις αρχές, το άρθρο 68 για, τις για την ειδική στήριξη επιτρέπει στα κράτη-μέλη να διατηρήσουν τέτοια καθεστώτα στήριξης για συγκεκριμένες περιστάσεις. Διατηρώντας ή δημιουργώντας τέτοιες μορφές ε, συνδεδεμένης ε, ε, στήριξης, το άρθρο 68 ουσιαστικά αποκλίνει από, τη γενική, από τη γενική στοχοθέτηση του πυλώνα 1. Βεβαίως ο στόχος του δεν ήταν να δημιουργήσει την επανασύνδεση, αλλά να δώσει κάποιες κομμένες και ραμμένες λύσεις, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των συγκεκριμένων προβλημάτων. Γιατί ο κανονισμός λέει ότι οι παρεκκλήσεις παρέχονται πολύ περιορισμένα και σε συγκεκριμένα συγκεκριμένε περιστάσει. Το ε, ελεκτικό συνέδριο λοιπόν εξέτασε το κατά πόσο η εισαγωγή αυτού του καθεστώτο ε, από το 1968 ε, και η εφαρμογή του συνάδουν με τι αρχέ που αναφέρονται στην νομοθεσία. Αν ήταν δηλαδή απαραίτητε, αν ήταν σχετικέ με την νομοθεσία και αν, ήταν, αν υπήρξε επαρκέ σύστημα ελέγχου για, την, ε, ε, για τον έλεγχο της εφαρμογής του καθεστώτος. Το συνέδριο ε, βρήκε ότι αυτή η ειδική στήριξη που προβλέπεται από το άρθρο 68 ήταν ένας, μια σύνδεση κατακρεματισμένων 113 συγκεκριμένα μέτρων με έναν συνολικό προϋπολογισμό 6,4 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2010 έως 2013. Ο έλεγχο επίση διαπίστωσε ότι το πλαίσιο που δημιουργήθηκε για να, ενισχυθεί, για να ενισχυθούν οι στηρίξει του άρθρου 68 ήταν ε, ε, μόνο για συγκεκριμένε ε, και ορισμένε περιπτώσει και έτσι το άρθρο 68 συνάδει με τι αρχέ τη πλούστευση και τη αποσύνδεση. Αυτές οι διατάξεις όμως ε, θεώρησε το ελεγκτικό συνέδριο ότι ήταν ε, ανεπαρκής. Η Κομισιόν δεν μπορούσε να ελέγξει την ε, αιτιολόγηση αυτών των περιπτώσεων και τα κρατημέλη είχαν τεράστια διακριτική ευχέρεια. Η Κομισιόν δεν μπορούσε να λάβει νομικώς δεσμευτικές δράσεις και τα κράτη-μέλη ως μόνη υποχρέωση είχαν να κοινοποιούν στην Κομισιόν τις προθέσεις τους να υποβάλουν τέτοια είδους διάταξη ειδική στήριξη. Επίσης, θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχουν επαρκές ενδείξεις για ότι τα μέτρα που ε, εισήχθησαν ήταν πάντα απαραίτητα σχετικά με τις ανάγκες, ε, την αποτελεσματικότητα και το επίπεδο στήριξης που είχε τεθεί. Επιπλέον, ε, ήταν ανεπαρκείς οι στόχοι και οι δείκτες και αυτό ε, θα εμποδίσει μάλλον την μελλοντική αξιολόγηση των συνεπειών αυτών των μέτρων. Τέλος, το ελεκτικό συνέδριο είδε κάποιες αδυναμίες στους διοικητικούς ελέγχους και αυτές οι αδυναμίες ε, δεν καταγράφηκαν παρά τους ε, ελέγχους που έγιναν και που ήδη ήταν ιδιαίτερο έντονη, αλλά που κάποιε φορέ πρέπει να είναι ακόμη πιο περίπλοκοι έτσι ώστε να πληρούν τι προποθέσει που θέτουν οι κανονισμοί. Το ελεκτικό συνέδριο λοιπόν έκανε μια σειρά συστάσεων στην έκθεσή του και θα, το θα τις επαναλάβω. Καταρχάς, η ειδική στήριξη για κάποιες ε, γεωργικές δραστηριότητες θα πρέπει να βασίζεται σε σωστή, αυστηρή ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 68 και η απόδοση αυτής της στήριξης θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς στην Κομισιόν και να ελέγχεται από αυτήν. Επίσης, για να μπορέσουμε να υποθέσουμε, για να μπορέσει μάλλον να αναλάβει την ε, ε, ευθύνη που έχει ε, η Κομισιόν στα πλαίσια της κοινή διαχείρισης, θα πρέπει να παίξει ένα πιο ενεργό ρόλο, θέτοντας τα κριτήρια που θα διέπουν την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Τρίτον, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δείξουν ότι κάθε ειδικό μέτρο στήριξης που θέλουν να εισαγάγουν είναι απαραίτητο ε, σε ό,τι αφορά την ανάγκη και την προσθέμενη αξία που θα φέρει με βάση τις ε, ε, παρακλήσεις. Είναι σχετικό σε σχέση με τις, με τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή, τα κριτήρια και τα επίπεδα στήριξης και ότι ικανοποιεί τα κριτήρια της χρηστής οικονομικής διαχείρισης. Τέλος, το Συμβούλιο, ε, το Συνέδριο, ε, είπε ότι εφόσον έχουν εισαχθεί κάποια μέτρα από τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να υπάρξει ε, η σωστή και συνολική διαχείριση και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξουν ελεγκτικά και εποπτικά συστήματα. Για να μην υπάρξει δυσχερές κόστος, το κράτος μέλος θα πρέπει να λάβει υπόψη και τους ελέγχους που έχουν γίνει στην όλη φάση σχεδιασμού ε, στα πλαίσια πάντα της ε, ε, απλούστευσης της, του ελέγχου των κριτηρίων κτλ. Ή ακόμη και στην απόφαση που έχει πάρει το κράτος μέλος να μην εφαρμόσει ένα τέτοιο μέτρο. Στη νέα κοινή γεωργική πολιτική Αυτή η ιδέα, αυτή η άποψη της ε, ειδική στήριξης ε, προβλέπεται από το άρθρο 68 και αντικαθίσταται από την εθελοντική, εθελούσια ε, συνδεδεμένη στήριξη που ορίζεται στα άρθρα 52-55 του νέου κανονισμού 1307 του 2013. Βεβαίως, τα μέτρα, παρόλο που τα μέτρα σε πρώτη ανάγνωση είναι περιορισμένα, έχει δοθεί μεγάλη διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη. Και όταν υιοθετήθηκε η έκθεση, Λέγεται στο, στο κείμενο ότι ο κατάλογος των προϊόντων και του ε, ορίου του προπολογισμού που είναι διαθέσιμο για τέτοια συγκεκριμένη στήριξη θα αυξηθεί και οι προϋποθέσεις για στήριξη θα εξαρτηθούν από την ε, ε ερμηνεία που θα δοθεί στο μέλλον σε πολύ ε, ασαφείς έννοιες όπως ε, δυσκολίες, ειδικό συμφέρον οικονομικό, για οικονομικούς ή ε, περιβαλλοντικούς σκοπούς ε, και τα περισσότερα συνδεδεμένα μέτρα στήριξης που υπάρχουν μπορεί να παραμείνουν. Η Κομισιόν ε, απήντησε ότι ε, σύμφωνα και με, τις, ε, με τα όσα έχει ορίσει η Κομισιόν είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους μέλους να ορίσει συγκεκριμένους τύπους καλλιέργειας ή γεωργικούς τομείς που αντιμετωπίζουν κάποιες ειδικές δυσκολίες και πρέπει να στηριχθούν. Γι' αυτό η εφαρμογή των μέτρων αυτών θα παραμείνει στη δικρατική ευχαίρεια των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά η Κομισιόν έχει καταδείξει ότι όλη αυτή η ιδέα των δυσκολιών θα οριστεί μέσω ε, συμπράξεων. Το ελεκτικό συνέδριο περιμένει να δει πώς θα ε, οριστεί αυτός ο όρος τελικά μέσω των κατεξουδότων συμπράξεων. Οπότε το Ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι σε αυτό το πλαίσιο και υπό το φως ε, της, ε, του σχεδιασμού του μελλοντικού εφαρμοστικού κανονισμού από την Κομισιόν, οι συστάσεις που εκφράζει το Ελεκτικό συνέδριο παραμένουν ενισχύ και βεβαίως θα, παραμένουμε, θα περιμένουμε να δούμε τις τελικές κατεξοδότητες συμπράξεις όταν αυτές υιοθετηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ και βεβαίως και εγώ και ο συνάδελφος είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε ερωτήσεις αν έχετε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα στην εισηγήτρια το λόγο. οκ. Βρω Κάντεμπαχ. Η κυρία Κάντεμπαχ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω το ελεκτικό συνέδριο. Το εκτιμούμε ε, που παρόλο που δεν είναι οι ελεγκτέ παρόντε εδώ, μπόρεσε να μα κάνει μια μικρή παρουσίαση. Δεν έχω να προσθέσω εγώ πολλά. Ε, βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση όπου έχουμε μια σειρά συστάσεων από το ελεκτικό συνέδριο, οι οποίες ε, θα πρέπει να εισρέψουν στη νέα κυριακή πολιτική, γιατί πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της κοινή πολιτική. πολιτικής. Είδαμε ότι υπήρχαν 113 διαφορετικά μέτρα. Ε, προφανώς η συγκρισιμότητα μεταξύ τους ε, είναι πάρα πολύ, η σύγκριση μεταξύ τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και βεβαίως κανένας δεν ξέρει και ποια είναι αυτή η επιπλέον χρήση ε, των ε, χρημάτων των φορολογουμένων και βεβαίω και για τα κρατημέλη ε, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το ε, ορίσουν. Ειδικά όταν μιλούμε για δυσκολίε κάτω από τις οποίες εμπίπτουν όλα αυτά τα περίπλοκα και διαφορετικά μέτρα που προβλέπονται. Η προβληματική αυτή λοιπόν που φαίνεται εδώ είναι ότι Γενικώ ε, στο κοινό είναι πολύ δύσκολο να παρουσιαστούν αυτά τα επιχειρήματα όταν δεν μπορούμε από την άλλη να αποδείξουμε και το, την ανάγκη, την χρησιμότητα αυτών των μέτρων. Αναφέρονται όλα αυτά στο άρθρο 52-55, παρόλο που ο, ο αυτός είναι πάρα πολύ ευρύς και πολύ γενικόλογος, θα πρέπει να περιμένουμε τις κατεξοδότητε συμπράξει τη Κομισιόν. Ελπίζω όμω ότι και η δική μου γνωμοδότηση, η γνωμοδότηση τη Επιτροπής μα εν πάση περιπτώσει, του Κοινοβουλίου, αλλά και οι ε, συστάσει ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου θα ληφθούν υπόψη από την Κομισιόν, γιατί δεν μπορεί η Κομισιόν να έχει στόχο μέσω τη ε, παραγράφου 55 να απορρίπτει αυτέ τι συστάσει. Θα πρέπει από την αρχή τα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν αυτές τις ε, συνδεδεμένες, ε, αυτό το καθεστώς συνδεδεμένων ε, στηρίξεων να ζητά επαρκείς αποδείξεις και επαρκή αιτιολόγηση. Αυτά και ευχαριστώ. Εύα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και το ανεκτικό συνέδριο. Κάποια από τα ζητήματα έχουν, είναι συνεκτικά, αλλά το πλαίσιο του άρθρου 68 και σίγουρα με την διακριτική ευχαίρεια που χορηγείται τα κρατη είναι απόλυτα σύμφωνα με την νομιμότητα. και αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία αυτή η στήριξη είναι ε, σύμφωνη με τις, ε, την ε, ενίσχυση. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε ειδικέ περιστάσει, ε, τομεί που αντιμετωπίζουν ε, οικονομικέ ή ε, περιβαλλοντικά προβλήματα. Φυσικά η διασυνδεμένη ενίσχυση επιτρέπει να αντιμετωπιστούν σημαντικά ζητήματα τα οποία δεν επιλύουν όμως, δεν μπορούν να φέρουν λύση του προβλήματο μέσω άλλου μηχανισμού. Το θέμα της μετέθυνσης του ΚΑΠ, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχαν στενές και εντατικέ διαπραγματεύσεις για τροποποίηση του άρθρου 68. Το αποτέλεσμα τη διαπραγμάτευση ήταν ένα νέο σχήμα, πολύ πιο διαφανέ, το οποίο θα επιτρέψει να, ε, ε, να αποδεχθεί η επικάλυψη με άλλα θέματα όπως αυτά της περιβαλλοντικής, ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν συνομοθέτης και μεγάλος υποστηρικτής των συνεδεμένων ενισχύσεων και των θέματων άμεσων πληρωμών που έχει τύχει διαπραγμάτευση μειώνει σημαντικά την γραμμή χρηματοδότηση που θα επηρεάσει του τομεί που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αυτή η κατάσταση λοιπόν μα επέτρεψε να να ωφελήσουμε τους ε, δικαιούχους Εξάλλου, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ευρωπή οι απαντήσεις που δίνονται από το, Ευρωπαϊκό, Συνέδριο ε, θα πρέπει να ενημερώσουμε περαιτέρω των Κομισιόν τους επιλεγέντες τομείς και τους λόγους για τους οποίους θέλει να χορηγήσει τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Ο εκ θα ήθελα να αναφέρω ότι καταλήξαμε σε μια συμφωνία ανάμεσα στα κοινωτικά όργανα και μαζί με το Κοινοβούλιο θα πρέπει να στηρίξουμε αυτό το συμβασμό, ο οποίο αναφέρει την ανάγκη αντιμετώπισης των δυσκολιών που με άλλο τρόπο δεν θα ήταν δυνατόν να ε, εφαρμοστεί. Φυσικά υπάρχουν κάποιες ελλείψεις ε, στον τομέα όπως συμβαίνει σε, σε όλη την ΚΑΠ γενικότερα. Αλλά η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από την Κομισιόν θα επιτρέψει να ε, χορηγηθούν, να, δίνουν, να δοθούν κυρώσεις ε, στα κράτη τα οποία έχουν παραβεί τους κανόνες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Το ελεκτικό συνέδριο θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ να πω πως ε, για μας ε, σημασία έχει να ενημερώσουμε και να προειδοποιήσουμε τους νομοθέτες σχετικά με τον περιοριστικό χαρακτήρα των μέτρων όπως είχε προβλεφθεί. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό στη μελλοντική ΚΑΠ και οι διατάξεις ε, τις οποίες ανέφερε το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου ε, να εφαρμοστούν σωστά, τόσο το καλύτερο, αλλά ε, θα πρέπει να αποδειχθεί κατά την διαδικασία αυτό. Ευχαριστώ. Και εγώ έκανα, ξέρετε, ένα μικρό λάθος. Θα έπρεπε να δώσω το λόγο και στον ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Παρακαλώ, ε, ε, πείτε μας και το όνομά γιατί δεν έχω κατάλογο παρόντων. Ευχαριστώ. Λέγομαι Φλάβιο Κοτούνη. Είμαι τμήματάρχης στη Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Ευχαριστώ λοιπόν για τη δυνατότητα ανταλλαγή απόψεων για αυτή την ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για τα ειδικά μέτρα στήριξη που χορηγείται με βάση το άρθρο 86 του κανονισμού 73 Ευχαριστώ τον Ελεκτικό Συνέδριο και την κυρία Κάντεμπαχ για τις παρατηρήσεις τους και τις συστάσεις τους. Κατά την περίοδο 10-13, 25 κράτη-μέλη αποφάσισαν να αξιοποιήσουν την ειδική βοήθεια με το άρθρο, βάσει του άρθρου 68. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εφαρμογή του σχέδιου ειδικών ενισχύσεων, ειδικών στηρίξεων, που χωρίζει δυνατότητα συνδεδεμένων πληρωμών, δεν θέτει να αμφιβόλω τη γενική κατεύθυνση των ε, απευθέων ενισχύσεων που είναι αποσύνδεση. Είναι, περιορίζεται στο 3,5% του εθνικού επίπεδου ενισχύσεων και είναι συμβατό με τις προδιαγραφές του ΠΟΕ, διότι στόχος είναι να διατηρηθεί το τρέχον επίπεδο παραγωγής και όχι να αυξηθεί οι συστάσεις του συνεδρίου κυρίως αφορούν τα κράτη-μέλη. Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίσουν ε, τους τομείς παραγωγής και τα είδη εκμεταλλεύσεων που μπορούν να υπαχθούν στο άρθρο 68. Τα κράτη-μέλη θεωρείται ότι είναι τα πλέον κατάλληλα για να καθορίσουν τις προτεραιότητες ανάμεσα στα διάφορα είδη στοχευμένης στήριξης και να καθορίσουν και τις περιοχές και τους κλάδους που έχουν τις περισσότερες δυσχέρειες. Παρόλα αυτά, έχουμε πλήρη συνέστηση ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες που αναφέρθηκαν και εδώ και έχουμε προτείνει και οι συνομοθέτες ενέκριναν ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής για το μέλλον. Μαζί με τα κράτη-μέλη η Επιτροπή θα κάνει τα αναγκαία βήματα για να εφαρμοστούν ε, τα μελλοντικά μέτρα μέσω και της ε, ε, προτινόμενης εθελοντικής συνδεδεμένης στήριξης, για παράδειγμα. Προτείνεται ένας κατάλογος των τομέων και παραγωγών, περισσότερη διευκρίνηση και να υπάρχει ανώτατο όριο για τις εθνικές ενισχύσεις ετήσια ανώτατα ώρα για αυτές τις ενισχύσεις και η έγκριση για την, από την Κομισιόν να είναι αναγκαία εάν προτίθενται τα κράτη-μέλη να υπερβούν το όριο. Εάν αποφασίσουν τα κράτη-μέλη να το εφαρμόσουν, πρέπει να ενημερώσουν την Κομισιόν για τους τύπους εκμετάλλευσης και τους τομείς και το επίπεδο στήριξης που προτίθενται να χορηγήσουν. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να αναφέρουν και τους λόγους για τους οποίους θέλουν αυτήν την συνδεδεμένη στήριξη και τι αποτελέσματα θέλουν να επιτύχουν. Όπου οι αποθάσεις των κρατών μελών απαιτούν υπέρβαση του συγκεκριμένου ποσοστού του εθνικού ανωτάτου ορίου, που είναι 8%, θα πρέπει να δοθεί αναλυτική πληροφόρηση για τον τομέα και την περιφέρεια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους εκμετάλλευσης ή κλάδου που απαιτούνται για να αυξηθεί για να δικαιολογηθεί η αύξηση της στήριξης. Και αν η αποφάση των κρατών μελών πρέπει να εγκριθεί, τότε θα πρέπει να υπάρχει λόγηση, για παράδειγμα, η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων ή η ανάγκη να ε, δοθεί ε, η αναγκαία πρώτη ύλη σε τοπικές μεταπητικές βιομηχανίες. ή προτάσεις για το 2013 της κοινή γεωρικής πολιτικής ε, περιλαμβάνουν και ένα πλαίσιο αποτίμησης και αξιολόγησης για να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των μέτρων και του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα της κοινή γεωρικής πολιτικής. Νομίζουμε ότι τα μέτρα αυτά θα βελτιώσουν την εφαρμογή του συγκεκριμένου αυτού μέτρου για να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες δυσχέρειες. Όπως είπαμε, ε, θα αναπτυχθεί περαιτέρω η εφαρμογή του μέτρου αυτού μέσω κατεξοδότηση πράξεων που συζητιούνται σε αυτή τη φάση. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. και με συγχωρείτε που δεν σας έδωσα απευθεία το λόγο. Κυρία Κάντεμπαχ, θέλετε να κάνετε τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου μπορούμε να συμπληρώσουμε την έκθεση. Αν έχετε άλλα αιτήματα, παρακαλώ, να μου τα αποστείλετε και ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ. Οπότε, λίγη και η εξέταση αυτού του θέματος και έχουμε την συνεδρίαση τώρα των συντονιστών. Αλλά πριν να, να πω κάτι προσωπικό στον Σέρεν Σέντεγκαρτ γιατί άκουσα ότι ο Σέρεν θα παραιτηθεί από το Κοινοβούλιο αποφάσισε να παίξει σημαντικό ρόλο περαιτέρω στην εθνική πολιτική της χώρας του της Δανίας. Άκουσα <clears throat> ότι είναι τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού όπου συμμετέχει ο συντονιστής της ΓΚΟΕ και από πλευράς άλλων συναδέλφων. Βέβαια δεν είναι πολύ παρόντες, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι εκφράζω την άποψη όλων λέγοντας ότι η συνεργασία ήταν ε, πολύ ευχάριστη με τον Σέρεν Αναλάβατε πολλές πρωτοβουλίες στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Ήσασταν πάντα επικοδομητικός. Είναι πραγματικά κρίμα που ε, φεύγετε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά σας εύχομαι για το μέλλον και για τα μελλοντικά σας καθήκοντα στο ε, Δανέσκο Κοινοβούλιο κάθε επιτυχία. Και παρακαλώ να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Για 11 χρόνια ήμουν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, έχω διατελέσει ευρωβουλευτής για σχεδόν δύο θητείες. Ε, προτίθεμαι να ξανακατεύω υποψήφιος για το ε, κοινοβούλιο της χώρας μου. Δεν ε, παίρνει κανείς μόνος του πάντα τις αποφάσεις του για τα θέματα αυτά, παίζουν ρόλο και οι αποφάσεις του κόμματός μου, αλλά προσβλέπω στα καινούργια μου καθήκοντα ε, ήταν ε, με μεγάλη χαρά που ήμουν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, μου άρεσε πάρα πολύ η εργασία μου εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Υπολογισμού. Ορισμένε επιτροπέ είναι πολύ πολιτικέ και η συνεργασία μεταξύ πολιτικών ομάδων δεν είναι πάντα εύκολη. Σε άλλε επιτροπέ που είναι πιο τεχνική δουλειά μπορεί να ασχοληθεί κανεί με συγκεκριμένα θέματα και πιστεύω ότι στην Επιτροπή μα παρά τι πολιτικέ μα διαφορέ και διαφορετικέ αφετηρίε πάντα κατορθώσαμε να συμφωνήσουμε ότι ε, τα χρήματα του φορολογουμένου πρέπει να δαπανώνται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Όλοι επιχειρήσαμε να συμβάλλουμε στην ε, επίτευξη αυτού του στόχου. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά. Σα ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνεργασία. Και θα θυμάμαι πάντα την συμμετοχή μας σε αυτήν την επιτροπή με μεγάλη χαρά. Εύχομαι σε όλου ό,τι καλύτερο. Σε όσου πρόκειται να ξανακατέμψουν εκλογέ, εύχομαι επίση καλή επιτυχία.